Uh, good morning, colleagues. Good morning, Mr. Brons. I think we were the only ones who were here at nine. Καλημέρα, συνάδελφε. Συνάδελφοι, κύριε Μπρόντς, ήσασταν ο μόνος που ήρθε εδώ από τις 9 μας με μένα. Okay. Can I ask everybody to take their... Καθίστε παρακαλώ ή τουλάχιστον ελάτε ήσυχα για να αρχίσει η συνεδρίαση. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 23 νέες ψυχοτρόπες ουσίες και ελάχιστες διατάξεις για τα συστατικά ε, στοιχεία και τις ελάχιστες ποινικέ κυρώσεις όσον αφορά την διακίνηση παράνομων ναρκωτικών ουσιών. Οι συγητές είναι ο κύριος Ποτασιέβιτς από το ΕΛΚ και ο κύριος Χιμένας Πεσερίλ επίσης από το ΕΛΚ. Ο κύριος Ποτασιέβιτς απουσιάζει σήμερα. Η παρουσίαση λοιπόν της έκθεσης θα γίνει από τον κύριο Λίσεκ. Το Νοέμβριο έγινε μια πρώτη παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο έκθεσης τώρα βρίσκεται ενώπιόν σας. Κύριε Λίσεκ, μπορείτε να παρουσιάσετε λοιπόν το κείμενο του κύριου Ποτασιέβιτς. Έχετε το λόγο. much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να στήσω συγγνώμη εκ μέρου του κυρίου Ποτασιέβιτ, ο οποίο ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Δυστυχώς, ευτυχώ υπάρχει μια συνεδρίαση του ε, Σχετικού Συμβουλίου που θα αποφασίσει τον κατάλογο των υποψήφιων για τι επόμενε ευρωεκλογέ. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική συνεδρίαση. Γι' αυτό και απουσιάζει ο κύριος Ποτασιέβιτ. Έπειτα, ε, να πω ότι χαίρομαι πολύ που πρώτη φορά μιλώ ενώπιον τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα παρουσιάσω λοιπόν τα κυριότερα σημεία και σχόλια του κυρίου Ποτασιέβιτς. Ο κύριος Ποτασιέβιτς καλωσορίζει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καν πρόταση κανονισμού που θα αποσύρει από την αγορά τις πιο επικίνδυνες ψυχοτρόπες ουσίες. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, το φαινόμενο αυτό των ψυχότροπων ουσιών οι οποίες είναι διαθέσιμες σε χώρες τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχετικά καινούριο. Η κατανάλωση όμως αυξάνεται με ταχύτητα τους και αποτελεί ένα πρόβλημα. Ορισμένες από αυτές τις ουσίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Ο εισηγητής θεωρεί ότι ο κανονισμός αυτός θα ελαχιστοποιήσει και ενδεχομένως θα βοηθήσει να ε, απαλληφθούν ορισμένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που προκαλούν οι ουσίες αυτά στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ε, λήψη αποφάσεων καθώς και μια ταχύτατη διαδικασία όσον αφορά την ταξινόμηση του επίπεδου κινδύνου που θα δώσει προστιθέμενη αξία στον κανονισμό. Ο παρόν μηχανισμός προβλέπει η διαδικασία για τις επικίνδυνες ε, ψυχότροπες ουσίες να είναι χρονοβόρος. Και αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να δράσουμε γρήγορα έτσι ώστε να παρέχουμε στους πολίτες μας τη μέγιστη δυνατότητα ασφαλείας. Έχουμε πάνω από 300 νέες ψυχοτροπές ουσίες που χρησιμοποιούνται και κυκλοφορούν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμφανίζονται με ρυθμό μία νέα ουσία την εβδομάδα. Η ταξινόμηση λοιπόν των ουσιών, ανάλογα με τον κίνδυνο που προκαλούν, ε, προβλέπεται να είναι ε, χαμηλή, μέτρια και μέτρια προς υψηλή και υψηλή. Ο κύριος Ποτασιέβιτς πιστεύει ότι ο κανονισμός αυτός ε, θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός ε, στα εθνικά μέτρα και στις τροπολογίες του αναφέρεται στο άρθρο 11 και το άρθρο 12 για τις ε, ουσίες χαμηλού και μέτριου κινδύνου. Σύμφωνα με τις ε, διατάξεις του κανονισμού δεν προβλέπεται καμία δράση για τις ε, ουσίες χαμηλού κινδύνου. Ο εισηγητής όμως πιστεύει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν περιορισμούς ή να εισαγάγουν νέους περιορισμούς για ε, νέες ουσίες. Αν αυτές προκα... έχουν... είναι αρκετά επικίνδυνες για την εκάστοτε χώρα. Οι ουσίες αυτές λοιπόν σε περίπτωση που χαρακτηριστούν ως ε, επικίνδυνες θα αποσυρθούν από την αγορά για να μην είναι προσβάσιμες στους καταναλωτές. Επίσης προβλέπονται μέτρα ελέγχου της κυκλοφορίας των ουσιών αυτών μόνο για συγκεκριμένους λόγους κατόπιν άδειας, όπως για παράδειγμα για την παρασκευή φαρμάκων. Ο κύριος Ποτασιέβιτς στην ε, έκθεσή του ζητά από τα κράτη-μέλη να λάβουν τα ίδια πρόσθετα μέτρα. Επίση, ο εισηγητή καλωσορίζει τι προσωρινέ ε, απαγορεύσεις και του προσωρινού περιορισμού στην αγορά για διάστημα 9 μηνών. Ε, οι περιορισμοί αυτοί θα επιτρέψουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρουν από την αγορά ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες με ε, ταχύτητα τους ρυθμούς εάν παρατηρηθούν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών ακόμα και σε ένα κράτος μέλος. Μια προσωρινή απαγόρευση των ουσιών αυτών θα εισηχθεί προτού γίνει η εκτίμηση και η ανάλυση των ουσιών αυτών και προτού εφαρμοστούν πιο μόνιμα μέτρα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ο κ. Ποτασιέβιτς πιστεύει ότι χρειάζεται οι ουσίες αυτές να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιστρέψουν ξανά στην αγορά. Γι' αυτό στην έκθεσή του προτείνει να δοθεί η δυνατότητα παράτασης της ε, απαγόρευσης για 12 επιπλέον μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και εξέτασης εφόσον η αξιολόγηση αυτή χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Ο κύριος ποτασιέβιτς στην έκθεσή του επίσης τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη για γρήγορη ανταλλαγή των ε, διαθέσιμων πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμακών. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ουσίες αυτές δεν προκαλούν μόνο για τον πολιτών αυτές καθ' αυτές, αλλά και ως συστατικό στοιχείο σε μείγματα άλλων ουσιών. Επίσης, ο συγητής τονίζει ότι για να είναι το σύστημα αποτελεσματικό χρειάζεται βελτιωμένος τρόπος συλλογής των ε, διαθέσιμων δεδομένων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και από όλους όσους έρχονται σε ε, επαφή και κάνουν αναλύσεις αυτών των ουσιών. Επίσης, ο εισηγητής τονίζει ότι βρισκόμαστε σε περίοδο λιτότητας και χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε υπόψη τους ε, περιορισμούς που έχουμε όσον αφορά τις ε, δαπάνες. Και πρέπει να δοθούν δυνατότητες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για πρόσθετους πόρους. Ο εισηγητής τέλος θα χαρεί πολύ να συνεργαστεί με τους κοιόδες εισηγητέ και με όλους ε, όσους ενδιαφέρονται για την έκθεση έτσι ώστε ο κανονισμός να υιοθετηθεί το γρηγορότερο δυνατόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χιμένες, έχετε το λόγο για τη δική σας έκθεση. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση να διευρύνει το πεδίο εφαρμογή της απόφασης του 2004 απόφαση πλαίσιο για τις ψυχότροπες ουσίες που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Προτασιέβης που είναι ο εισηγητής για τον κανονισμό για το ίδιο θέμα και με αυτόν ήταν πάρα πολύ εργαστή συνεργασία. Πρόκειται για κάποια... Πρόκειται για αυτές αυτά τα ναρκωτικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ε, ζημιά ή στην ε, υγεία και την ε, ασφάλεια. Πρόκειται για μεγάλο βάρος για την κοινωνία και αυτό έχει να κάνει με τη λειτουργία του εγκεφάλου και επίσης σαν συμπτώματα έχουμε την αλλίωση της συνείδησης, της συμπεριφοράς κλπ. Ε, οπότε όλα αυτά ε, έχουν απασχολήσει το παρατηρητή ναρκωτικών και ε, τοξικομανίας. έχουν συνεργαστεί το Κοινοβούλιο με Κομισιόν και κράτη-μέλη. Και αυτό το οποίο επετέφθη είναι ότι από πλευρά Ένωση είπαμε ότι θα πρέπει να επισημάνουμε το ότι αυτές οι νέε είναι πηγή ανησυχίας, πηγή κινδύνου για την υγεία των Ευρωπαίων. Πάρα αυτά να μην υποτιμήσουμε το έργο της καταπολέμησης, της διάδοσης, της διανομής αυτών των ε, ουσιών. Πρόκειται για μια αγορά διαδικτυακή που πάρα πολύ γρήγορα ε, γίνονται αλλαγές ε, επαναστατικές όσον αφορά την, τις πωλήσει κλπ. Οπότε αυτοί που κατασκευάζουν αυτές τις ουσίες ανταποκρίθηκαν στο κοινό νομικό πλαίσιο και με νέους μηχανισμούς τα θέτουν αυτές τις ουσίες στην εμπόρια, έχουν διάφορους διάβλους ε, νομιμοφανείς και επίσης έχουν αλλάξει την μοριακή δομή των ουσιών αυτών και οπότε έτσι παρακάμπτουν τον νόμο χωρίς να αλλάξουν τα αποτελέσματα τα οποία επιφέρουν αυτές οι ουσίες στους χρήστες τους. Επίσης, ε, αυτές οι ουσίες τώρα ξεφεύγουν από τον νόμο πολύ πιο εύκολα από ό,τι τα κλασικά ναρκωτικά. Επομένως τώρα βλέπουμε ότι χρειάζεται πιο δραστήρια ε, πολιτική πλευρά των ε, κρατών μελών, ώστε οι γενεί κίνδυνοι να αντιμετωπιστούν. Οπότε έχουμε την τροπολογία υπερθμών 5 και την τροπολογία υπερθμών 6. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να παράσχουν κάποια δεδομένα όσον αφορά το πώ ε, κατασκευάζονται αυτά τα ναρκωτικά, ποια είναι τα εγκλήματα τα σχετιζόμενα με την πώληση αυτών των ναρκωτικών, το ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η πώληση ε, στους ανηλίκους και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν αναλύσεις ε, των ναρκωτικών αυτών και βέβαια θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε τους διάφορους κινδύνους γιατί το παρατηρητή τα ναρκωτικά ε, κατέληξε στο ότι αυτά τα προϊόντα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και επομένως προτείνει την απόσυρση από την αγορά. Έχουμε μια προθεσμία 12 μήνη, οπότε και μετά τους 12 μήνες θα υπάρξουν κυρώσεις σε όσους θέτουν σε εμπορία και κυκλοφορία τέτοια ναρκωτικά στα κρατημέλη. Επίσης τονίζουμε το ότι εύκολα μπορούν τα κρατημέλη να εφαρμόσουν ε, ε, αυτό, αυτή την νομοθεσία μέσα σε αυτό το 12 μήνο. Έχουμε την τροπολογία υπαριθμών 3 και εκεί λέει ως διατύπωση τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τις διατάξεις της αποφάσεις πλαίσιο του 2004 το πιο σύντομο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 12 μήνες θα πρέπει να ενεργήσουν ταχαίως και ε, θα, έχουμε, ε, θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν και η παραγωγή αυτών των ουσιών, ή αλλιώ πρέπει να υποστούν τι κυρώσει του νόμου για αυτέ τι ψυχοδοσίε και τέλο πάντων τα συμπτώματα αυτών των, των ουσιών εκδηλώνονται όταν αυτέ οι ουσίε καταναλώνονται ε, μαζί με κάποιε άλλε ουσίε που αναφέρονται σε έναν κατάλογο. Και υπάρχει ο σχετικό ορισμό αυτών των ενιών και επίση εξαθαρίζουμε ότι σε αυτή την οδηγία δεν ε, περιγράφεται ω έγκλημα η κατοχή αυτών των νέων ψυχοτρόπων ουσιών για προσωπική χρήση περιμένω πώς και πώς να συνεργαστώ με τους ε, υπόλοιπους ε, εισηγητές και να τροποποιήσουμε έτσι το κείμενό μας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας προτείνω τώρα να ακούσουμε πρώτα τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Προεδρία του Συμβουλίου και κατόπιν να αρχίσει η συζήτηση. Ε, μέχρι τώρα έχει ζητήσει ένα συνέντευξο το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρία Σπινόντα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ καταρχήν τους δύο εισηγητές, τον κύριο Ποτασίεβιτς και την κυρία Χιμένεθ, για την πολύ επικοδομητική δουλειά που κάνανε πάνω σε αυτό το πολύ στέρεο σχέδιο έκθεσης που μας υπέβαλαν. Και οι δύο εκθέσεις βλέπουν πολύ καλά το πρόβλημα που δημιουργούν οι νέες ψυχότροπες ουσίες, το πόσο περίπλοκες είναι και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης για να δώσει απαντήσεις ε, στα προβλήματα. Γιατί έχουμε να κάνουμε μια αγορά περίπλοκη, νέες ουσίες εμφανίζονται κάθε εβδομάδα, εξαπλώνονται πολύ γρήγορα και δημιουργούν διαφορετικούς κινδύνους κάθε φορά. Και τα δύο σχέδια έκθεσης τονίζουν και προσπαθούν να ενισχύσουν περαιτέρω τα βασικά σημεία της προστιθέμενης αξίας της πρότασής μας. Σας παραμπέμπω στο γεγονός ότι οι προτάσεις θα εξασφαλίσουν πιο αποτελεσματική δράση στις νέες ψυχότροπες ουσίες, επιτρέποντας και μέτρα περιοριστικά να μπουν πολύ νωρίτερα ε, στη διαδικασία μέσω προσωρινών μέτρων, αλλά και να συνοδεύσουμε τα εθνικά μέτρα για τις ουσίες αυτές. Οι προτάσεις τροπολογιών που κάνουν οι συγητές πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση να ενισχύσουν την προστιθέμενη αυτή αξία. Επίσης, η έκθεση ενισχύει περαιτέρω την πρόταση της Κομισιόν για πιο αναλογική δράση στις νέες αυτές ουσίες. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο προστιθέμενης αξίας. Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ε, μια προσέγγιση με περισσότερες αποχρώσεις. Οι δράσεις για τις νέες ουσίες θα εξαρτάται και θα είναι αναλογική ως προς το επίπεδο του κινδύνου. Γιατί, Γιατί πιστεύουμε ότι πιο επιβλαβείς ψυχότροπες ουσίες ε, που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο θα πρέπει να, να καλυφθούν από το ποινικό δίκαιο, οι υπόλοιπε από το διοικητικό δίκαιο. Αυτή η αναλογική προσέγγιση θα εξασφαλίσει καλύτερη προστασία των θεμητών χρηστών των νέων αυτών ουσιών, γιατί πολλές από αυτές τις ουσίες έχουν και άλλες χρήσεις, πέρα από το ότι χρησιμοποιούνται για, να, για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή φαρμάκων στη χημική βιομηχανία, στην βιομηχανία α, υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχουν τόσες πολλές ουσίες στην αγορά και είναι τόσο καινούργιες που είμαστε σε φάση έρευνα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι πιθανέ χρήσει. Επίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και την αξιολόγηση κινδύνου επί των ουσιών και οι τροπολογίε που προτείνουν οι δύο εισηγητέ ακριβώ ενισχύουν αυτό το τελευταίο στοιχείο. Συμπερασματικά. Καλωσορίζουμε και τι δύο εκθέσει. Εκτιμούμε τις βελτιώσεις που επιφέρουν και μεγάλη χαρά θα απαντήσουμε στις διαπραγματεύσεις ευελιξία για τα κράτη-μέλη να πάνε πιο πέρα από τα μέτρα που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαίρουμε τους συζητητές για το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση των εκθέσεων και ευχόμαστε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ καλή τύχη. Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις ε, μέσα σε αυτό το φιλόδοξο ε, χρονικό ορίζοντα. Από την Ελληνική Προεδρία, κυρία Ραπτάκη σε όλους από την Ελληνική Προεδρία. Ε, ε θα συνεχίσω στα αγγλικά. Ε, both the previous and the current president... Και η προηγούμενη Προεδρία και η σημερινή Προεδρία δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το φάκελο και θα δώσει στις συνεδριάσεις ομάδα εργασία την τέουσα σημασία. Ε, οι εμπειρογνώμονέ μα είναι το χώρο τη υγεία και την εφαρμογή του νόμου και θα εξετάσουμε όλες τις διατάξεις του σχεδίου πρότασης, ούτως ώστε να έχουμε το πιο αποτελεσματικό σύστημα για να αντιμετωπίσουμε τις νέες αυτές ψυχότροπες ουσίες που αποτελούν μεγάλη πρόκληση στις πολιτικές καταπολέμησης των ναρκωτικών και στην υγεία των πολιτών. Η συζήτηση στο Συμβούλιο για τον Κανονισμό ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2013 και το σχέδιο πρότασης συζητήθηκε στις τρει συνεδριάσεις επιληφωνικής προεδρίας. Επί ελληνικής προεδρίας η πρόταση για ένα κανονισμό ήδη έχει συζητηθεί στις 9 Ιανουαρίου φέτος στην οριζόντια ομάδα ναρκωτικών και η συζήτηση θα συνεχίσει και στις επόμενες συνεδριάσεις. Ε, έχουμε μάλιστα τρεις συνεδριάσεις το Φεβρουάριο για αυτό το θέμα. Η οριζόντια ομάδα ναρκωτικών με τους εμπειρογνώμονές της επικεντρώνει την προσοχή στα εξή θέματα τη νομική βάση της πρότασης, την επιλογή μεταξύ νομικής βάσης εσωτερικής αγοράς ή δημόσιας υγείας, ε, σύστημα αξιολόγησης κινδύνου, κριτήρια ε, και επίπεδα των κριτήριων που προβλέπονται, γιατί κάποιες αντιπροσωπείες μίλησαν για τις δυσκολίες συλλογής πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες ουσίες. Για τη δυνατότητα εισαγωγής εθνικών και πιο αυστηρών μέτρων σε σχέση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμούμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωράει γρήγορα, έχει ήδη προχωρήσει, βασιζόμαστε στη συνεργασία σας, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες νομοθετικές τροπολογίες που θα περάσουν έγκαιρα. Είναι για το καλό όλων να συμφωνήσουμε για τον κανονισμό, γιατί αυτό είναι προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη έχει στήσει το λόγο σχεδόν εισηγήτρια για τους σοσιαλδημοκράτες, κυρία Χέντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, δύο εισηγητές για το σχέδιο έκθεσης και να πω ότι στηρίζω την ε, γενική γραμμή που ακολουθούν. Ελπίζω με αυτή την έκθεση να αποκτήσουμε ένα κατάλληλο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε την ε, κυκλοφορία και την εισαγωγή αυτών των συνθετικών ναρκωτικών ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να θεωρηθεί ένα, ως ένα επιπρόσθετο μέτρο. Γι' αυτό λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα προστιθέμενη αξία του κανονισμού αυτού. Έχω ορισμένες ε, προτάσεις για τροπολογίε που θα υποβάλω και στου ε, συνεισηγητέ. Καταρχάς, η σύνδεση των ευρωπαϊκών με τα εθνικά μέτρα. Τι μπορούν οι αρχές των κρατών μελών να κάνουν όταν κάτι έχει ήδη γίνει σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια είναι τα πρόσθετα μέτρα που μπορούν να πάρουν τα κράτη-μέλη και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των τροπολογιών 15 και 16 στο σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα να μάθω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 15 και 16, τα οποία θα αλλάξουν την ε, δομή του κανονισμού με την εισαγωγή των τριών αυτών επιπέδων επικινδυνότητας. Επίσης, ε, ε, σε απάντηση στην κυρία Χιμένες να πω ότι στην πρόταση βλέπω ότι προβλέπονται εκτελεστικές πράξεις ποινικοποίηση των ουσιών αυτών. Δηλαδή στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να αποφασίσει για το τι θα αλλάξει και τι όχι. Θα ήθελα προσωπικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι εκείνο που θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις. Δεν ξέρω αν, έχουν, αν έχει ζητηθεί από τις νομικές υπηρεσίες να γνωμοδοτήσουν σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βέμπερ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση αυτή, η οποία μου φαίνεται αρκετά λογική και αναγκαία. έχει αυξηθεί η ζήτηση στην αγορά για τις νέες αυτές ε, ψυχοτροπές ουσίες. Το βλέπουμε αυτό και αυξάνεται η ζήτηση αυτή καθημερινά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές για τη δουλειά τους και την καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Νομίζω πως η πρόταση είναι λογική, διότι πραγματικά σκοπό έχει να προστατεύσει την αγορά με τους περιορισμούς αυτούς, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν η καλύτερη λύση είναι να παραταθεί το χρονικό διάστημα των περιορισμών μέχρι να γίνει η αξιολόγηση ή αυτή η αξιολόγηση να γίνει πιο γρήγορα. έτσι ώστε να αποτραπεί η κυκλοφορία των ουσιών αυτών στην εσωτερική αγορά. Εντάξει, υπάρχουν κάποια σημεία που μπορούμε να αλλάξουμε όσον αφορά την διατύπωση και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, αυτό που δεν θέλουμε είναι να ποινικοποιούνται οι χρήστες. Θέλουμε το αντίθετο, οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα θεραπείας. Γι' αυτό και θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες και να πω επίσης ότι η προσέγγιση μου φαίνεται πολύ καλή. Το να δοθεί δηλαδή στα κράτη-μέλη η δυνατότητα ευελιξίας όσον αφορά το πώς θα αντιμετωπίσουν τις ε, ουσίες αυτές. διότι τα τελευταία χρόνια ακολουθείται μια διαφορετική τακτική όσον αφορά τις ουσίες που ήδη χρησιμοποιούνται, που ήδη κυκλοφορούν. Ιδιαίτερα όταν αρχική πρόθεση για μια ουσία ήταν να χρησιμοποιηθεί για κάτι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό πιστεύω πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να ε, παρέχουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να ρυθμίζουν μόνα τους τις ουσίες αυτές. Ελπίζω πάντως να έχουμε ένα πολύ καλό νομοθετικό αποτέλεσμα, να έχουμε ένα νομοθέτημα το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες, θα είναι λογικό και ελπίζω να ολοκληρωθεί το έργο αυτό πριν τις επόμενες ευρωεκλογέ. Αυτό όμως εξαρτάται από τις ε, διαπραγματεύσεις, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Τελευταίος ε, ομιλητή στο καταλογό μου, ο κύριος Σλίτερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος για την σύνδεση αυτής τη πρότασης με τη λειτουργία του κανονισμού REACH. Διότι όταν μία ουσία έχει αφαιρεθεί από τον κανονισμό REACH είναι μια κάπως περίεργη διαδικασία. Καταρχάς πρέπει πρώτα να γίνει μια αναφορά από τα κράτη-μέλη. Μετά αυτό να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να γίνει αξιολόγηση και να βγει το τελικό πόρισμα. Για κάποιες άλλες ουσίες που δεν ξέρουμε ποιο αποτέλεσμα θα έχουν στους πολίτες, πρέπει να περιμένουμε πρώτα το τι θα γίνει και το τι θα αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εταιρείε παρασκευής φαρμάκων έχουν πολλές φορές κάνει ήδη εκ των προτέρων τη δική τους ε, αξιολόγηση και τις δικές τους μελέτες. Προσπαθούμε να απλοποιήσουμε κάτι για τα πιο επικίνδυνα προϊόντα, όμως πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές η πρόταση αυτή είναι αρκετά ε, χαλαρή αυτή η εκτίμηση, αυτή η αξιολόγηση που προτείνεται να γίνει από την Επιτροπή ήδη έχει γίνει από την ε, φαρμακοβιομηχανία, οπότε θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις σε αυτό και θα υποβάλω και τροπολογίες έτσι ώστε να συμπεριληφθεί αυτή η απέτηση οι εταιρείε παρασκευή των ουσιών αυτών έχουν κάνει πρώτα τη δική του αξιολόγηση προτού περάσει αυτό στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, με ανησυχεί το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που θα αποφασίζει αν μια ουσία είναι επικίνδυνη ή όχι. Παρομοίως και για το συνδυασμό ουσιών. Η πρόταση 619 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται σε αυτούς τους συνδυασμούς. Όμως έχει προσθεθεί και μία παράγραφος από τους εισηγητές, η οποία λέει ότι αν μία τέτοια ουσία είναι παρούσα σε έναν συνδυασμό, σε ένα μείγμα, ήδη καλύπτεται. Δεν ξέρω αν χρειάζεται λοιπόν κάποια πρόσθετη τροπολογία. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας το εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, με ανησυχεί αυτή η κατηγοριοποίηση των ουσιών. Αυτές οι ομάδες, οι νέοι αυτή τη στιγμή βρίσκουν μια νέα ουσία, την δοκιμάζουν, μετά την απαγορεύουμε, ύστερα αλλάζει η χημική της σύσταση κατά ένα μόριο, είναι σχεδόν η ίδια και πάλι κυκλοφορεί στην αγορά νόμιμα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν υπάρχει κάποια διάταξη, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς κάποια έτσι ώστε να στοχεύσουμε αυτές τις ε, ενεργές ομάδες των χημικών ουσιών, χημικές ε, ουσίες δηλαδή, οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία. Για παράδειγμα η κοβέινη και η κοκαίνη είναι παρόμοιες ουσίες. Έχουν διαφορετικές ε, επιδράσεις, όμως ένα μόριο χρειάζεται μόνο να αλλάξει. Μπορούμε λοιπόν να κατηγοριοποιήσουμε σε ομάδες με έξυπνο τρόπο αυτές τις ουσίες έτσι ώστε να μην μπορούν να παρακάμπτουν τον νόμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να πω στις Ευχαριστούμε κύριε Σλίτερ. Ο κύριος Λίσεκ από ό,τι βλέπω έχει φύγει. Κυρία Χιμένες, είστε εδώ. Θα θέλατε εσείς να απαντήσετε ή να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα να απαντήσει σε ερωτήσεις του κυρίου Σλίτερ. Ναι, να απαντήσω στην ερώτηση. Αλλά να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ο άλλος συνεισηγητής δεν παρίσταται εδώ που συνέταξε αυτό το σημείο του κειμένου. Αυτό που με ρωτήσατε για τις διατάξεις του νόμου δεν αφορούν τις δικές μου τροπολογίες, αλλά του άλλου συνεισηγητού. Πάντως, ζητήσαμε γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία. Ε, πριν τις 28 του μήνος θα την έχουμε. Οπότε και τότε στα σίγουρα θα σας πω. Όταν πάρουμε την γνωμοδότηση θα σας απαντήσουμε. Και συγκεκριμένα ο συνεισηγητής και οι συνεργάτες που θα σας πούνε. Τώρα. Γι' αυτό που είπε η κυρία Βέμπερ Έχουμε τις τροπολογίες 3, 5 και 6 εκεί που αναφέρονται τα κρατημέλια και σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να αποφασίσουν τα κρατημέλια από μόνα τους. Αλλού όμως πρέπει να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να αποφύγουμε την ποινικοποίηση του κατόχου της ουσίας. Οπότε με τη σχετική τροπολογία θα το διορθώσουμε αυτό το σημείο. Sí. Sí, yo creo que respecto al Rich prefiero que Α, για το Rich. Καλύτερα μας τα εξηγήσει η Επιτροπή. Ε, ευχαριστούμε λοιπόν. Μήπως μπορεί να μας ξεκαθαρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται. Τι ισχύει με το Rich, την οδηγία για τα χημικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτές τόσο εύστοχες ερωτήσεις των βουλευτών και με τη σειρά να απαντήσουμε. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά την ερώτηση της, της κυρίας Head για την ευελιξία των κρατών μελών, για τη σχέση μεταξύ των ε, μέτρων της Ένωσης και των εθνικών μέτρων. Πολύ σημαντικό. Σας τονίζω ότι εμείς αυτό το οποίο έχουμε προτείνει και έχουμε την απόφαση 387 του Συμβουλίου, τα κρατημέλη θα συνεχίσουν να έχουν την αρμοδιότητα για τις περισσότερες περιπτώσεις που αφορούν τις ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά. Από περίπου 300 ουσίες που έχουν κοινοποιηθεί από τα κρατημέλη από το 1997 μόνο σε 10 περιπτώσεις έχουν ληφθεί μέτρα σε επίπεδο ένωσης, διότι όλες οι άλλες ουσίες δεν θεωρήθηκε ότι σε επίπεδο ένωσης παρουσιάζουν πρόβλημα. Οπότε και θεωρούμε τα κράτη-μέλη είναι θέση καλύτερα να χειριστούν αυτό το θέμα σε εθνικό επίπεδο. Οπότε, σύμφωνα με τις προτάσεις μας, θα αναλυθεί δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης, άπαξ κάποια ουσία έχει επισημανθεί σε μια σειρά κρατών μέλων και έχει διαπιστωθεί ότι σε αυτά τα κράτη-μέλη δημιουργεί πρόβλημα. Επόμενε περισσότερε αποφάσει θα λαμβάνουν σε εθνικό επίπεδο τώρα όσον αφορά τι ουσίε για τι οποίε αναλαμβάνουμε δράση και για τι οποίε υπάρχουν κατασταλτικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη σύμφωνα με την πρότασή μα πρόκειται να είναι θέση να προχωρήσουν κι άλλο σε πιο αυστηρά μέτρα εάν επιθυμούν με κάποια συγκεκριμένη ουσία, διότι σε εθνικό επίπεδο έχει επισημανθεί μεγαλύτερο κίνδυνο γιατί πίν ε, μια ουσία χρησιμοποιείται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο από κάποιους συγκεκριμένους και υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος οπότε ε, η Γερχημένη μα είπε για αυτές τις τροπολογίε, 15, 16, 17 Οπότε έτσι διευκρινίζεται το τι ισχύει σε περίπτωση που έχουμε και ουσίε χαμηλού κινδύνου ή μέσου κινδύνου. Οπότε τα κρατημέλη σε αυτή την περίπτωση θα είναι στέση να λάβουν μέτρα ή να λάβουν μέτρα συμπληρωματικά των ε, κοινοτικών και θα κοινοποιούν το τι μέτρα λαμβάνουν με το συγκεκριμένο σύστημα κοινοποίηση. Και έτσι θα είναι η κατάσταση ξεκάθαρη, θα υπάρχει διαφάνεια και θα προστατευτεί η ιστορική αγορά. Τώρα, για το REACH, πάρα πολύ εύστοχη ερώτησή σας. Σύντομα σας απαντώ ότι το REACH δεν καλύπτει αυτές τις ουσίες. Μόνο κατά εξαίρεση. Σε περίπτωση που έχουμε κάποια ουσία που χρησιμοποιείται από την χημική βιομηχανία, όπως το GBL, και το χρησιμοποιούν για ψυχαγωγία ορισμένη ο περιορισμός ο ποσοτικός, δηλαδή για κάποιες ουσίες που κυκλοφορούν σε μικροσίες, δεν χρειάζεται να πρωτοκολληθούν, να καταχωριστούν, όπως απαιτεί το REACH. Όμως, αναφέρονται από το REACH. Πάντως η εξορία στο κίνδυνο σύμφωνα με το REACH δεν λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο του καταναλωτή από την χρήση αυτών των ουσιών. Όπως κατά τα λοιπά προβλέπει το Ριτς και οι δικές μας προτάσεις. Επομένως το Ριτς δεν καλύπτει αυτές τις ουσίες, αλλά έχουμε προτείνει να συνδεθεί περισσότερο αυτή η νομοθεσία με το Ριτς. και επίσης να εμπλακεί η υπηρεσία των χημικών, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία των Χημικών Ουσιών και έτσι να δούμε τι γίνεται με τους κινδύνους από αυτές τις ουσίες τώρα. Οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πριν θέσουν συμπορία με τέτοια ουσία. Επίσης έχουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο σύστημα θέση συμπορία ψυχοτρόπων ουσιών. Αλλά έχουμε ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο αυτές που οι ουσίε που ήδη κυκλοφορούν για κάποιες χρήσεις που υπάρχουν στην αγορά τέλος πάντων γιατί κάποιος τις κατασκεύασε και τις πουλάει σε κάποιο κατάστημα και έχουμε αυτό το σύστημα για να αξιολογεί το κίνδυνο των υπάρχουσών ουσιών και σήμερα αυτό το σύστημα επίσης μπορεί να αποσυρθούν από την αγορά ίδιες ουσίες οπότε δεν έχουμε άλλα κριτήρια θέσεις σε εμπορία ή κάποιες προϋποθέσεις για τους συναλλασσόμενους που θέλουν να ρίξουν στην αγορά κάποιες τέτοιες οπότε Κάτι άλλο για την κυρία Βέμπερ. Ναι, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν το δικό του σύστημα για αυτές τις ψυχοτροπές ουσίες. Έχουμε μια σειρά διαφορετικών συστημάτων. Ε, υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα σε κάθε κράτος και οπότε το ζήτημα είναι ότι εμείς θέλουμε τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δικών μας μέτρων και των εθνικών. Αλλά θέλει το λόγο, βλέπω, λέει ο πρόεδρος. Θέλει πάλι το λόγο κύριο Να μην αρχίσουμε τώρα με κουβέντα για το Ρίτς, να το αφήσουμε και να πάμε στο επόμενο θέμα της μέσης διάταξης. Μισό λεπτό μόνο. Πολύ σύντομη ερώτηση. Αλλιώς να πάτε να τους βρείτε μετά τη συνεδρίαση. Όχι, δεν θα σου πω για το Ρίτς, παρά το ότι με ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Για πέστε μου. Εάν κάτι προορίζεται για κατάποση ας πούμε μια τέτοια ουσία γιατί δεν έχουμε ε, το, δεν έχουμε το νομοθέτημα για τα τρόφιμα. Ναι, αλλά αυτές οι ουσίες δεν κατανοούνται μόνο με κατάποση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να πάρει κανείς αυτές τις ουσίες. Η κατάποση είναι μόνο ένας τρόπος. Ένας από τους τρόπους. Οπότε, ε, αν επικαλεστούμε κάποιο άλλο είδους νομοθεσία και όχι την νομοθεσία για τις ψυχότροπες, τότε δεν θα έχουμε συστηματική αντιμετώπιση, συστηματική αξιολόγηση και συστηματική απόσυρση από την αγορά. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Οπότε τέλειωσε αυτό το σημείο της διάταξης. Κύριε Γκόμες, μόλις μπήκε στην αίθουσα που είναι η επόμενη συγγήτρια. Έχουμε το επόμενο σημείο το οποίο είναι το εξής. Α, για τις τροπολογίες Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου, 12 ώρα το μεσημέρι, έχετε προθεσμία για τις τροπολογίες. Και για τις δύο εκθέσεις, Χιμένεθ και Ποτασίεβιτς. Συμφωνία τώρα πλαίσιο ε, εταιρική σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της, αφενός και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την επανεισδοχή. Η συγκίτρια είναι η κυρία Γκόμες. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για αυτό το σημείο στις 16 Δεκεμβρίου Ακούσαμε παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο που εξήγησαν το διαχωρισμό της συμφωνίας σε δύο διαφορετικές διαδικασίες. Θα ακούσουμε λοιπόν καταρχήν την κυρία Γκόμες. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Είναι σημαντικό οι βουλευτέ να γνωρίζουν ότι αυτή τη βδομάδα η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε την έκθεση για αυτή την ε, συμφωνία πλαίσιο εταιρική σχέση και συνεργασία με την Ινδονησία. Η Ινδονησία είναι μια πολύ σημαντική χώρα στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Είναι μια κεντρική χώρα στην ε, ΑΖΕΑΝ και έχει πάνω από 240 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι η τέταρτη πιο πολυπληθής ε, χώρα. Είναι πολύ νεαρή χώρα. Το 40% είναι κάτω των 25 χρονών, 45% των κατοίκων. Είναι δημοκρατία πλέον και είναι ενδιαφέρον γιατί είναι μια δημοκρατία όπου το 90% των ανθρώπων είναι μουσουλμάνοι και βρίσκεται σε αυτό το αρχιπέλαγος πάνω από 17.000, που έχει πάνω από 17.000 νησιά και, έχει, και απλώνεται από τον Ινδικό ως τον Ειρηνικό σε πάνω από 5.000 χιλιόμετρα. Είναι μια χώρα ε, διαμετακόμιση διέλευση. Όσοι θέλουν να φτάσουν στην Αυστραλία πρέπει να περάσουν από εκεί ή όσοι περνάνε, ξεκινάνε από την Νοτιοανατολική Ασία, επίσης περνάνε από εκεί. Όποιο μετακινείται στην Ασία ουσιαστικά περνάει από εκεί. Αυτή η συμφωνία λοιπόν εταιρική σχέση και συνεργασία που υπογράφτηκε το 2009 και επικυρώθηκε από όλα τα, ευρωπαϊκά, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το οποίο δίνει τη σύμφωνη γνώμη του το Κοινοβούλιο με βάση την ε, έκθεση της ΑΦΕΤ η οποία υφαντήθηκε και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Μαρτίου. Αυτή η συμφωνία λοιπόν τι προβλέπει. Μία ρήτρα επανεισδοχής στο άρθρο 34.3. Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη ασιατική χώρα που υπογράφει μια συμφωνία επανεισδοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να παρεμποδίσουμε και να ελέγξουμε την παράτυπη μετανάστευση και την άτυπη μετανάστευση. Και λέει ότι αυτό συνάδει με τις διεθνείς υποχρεώσεις και την αρχή της μη επαναπρόθεσης. Έχει λοιπόν αμοιβέ υποχρεώσει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ινδονησία να, επαν... να δέχονται πίσω του συμμεταπού του. Συνδέοντα αυτή την έκθεση για τη ΛΥΜΠΕ, θεώρησα ότι είναι σημαντικό να ζητήσουμε η Κομισιόν να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες τις φάσεις της Συμφωνίας Επανεισδοχής και για όλε ούτω ή άλλω τι συμφωνίε επανεισδοχή υπάρχει αυτό το αίτημα και για αυτήν προφανώ. Υπάρχει δυνατότητα αναστολή σε περίπτωση που τα θεμελιώδη δικαιώματα παραβιάζονται. Επομένω, συστήνω στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδονησία να αναπτύξουν μια πλήρη συμφωνία ε, επανεισδοχής. Γιατί τώρα έχουμε απλώς μια ρήτρα ε, για την επανεισδοχή και όχι μια συμφωνία 100% η ρήτρα αυτή είναι ενταγμένη, είναι ενταγμένη στη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία και θα ε, συμπεριλαμβάνει και του υπηκόου τρίτων χωρών και του απάτριδε. Είναι σημαντικό αυτό, διότι αυτή η χώρα είναι μεγάλη χώρα διέλευση για την παράτυπη μετανάστευση, όπω σα είπα. Φυσικά θα ήθελα αυτή η ρήτρα επανεισδοχής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδονησίας να λάβει την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Αλλά πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να δημιουργηθεί μια πλήρης συμφωνία επανεισδοχής, μια καθαυτό συμφωνία επανεισδοχής με την Ινδονησία, όχι απλώς μια ρήτρα επανεισδοχής. Ευχαριστώ. Κομισιόν και η Προεδρία θα ήθελα να σχολιάσουν και εν συνεχεία θα δώσω το λόγο σε ερωτήσεις και θα γίνει μια συζήτηση. Βλέπω βέβαια ότι δεν έχουμε πολλού ευρωβουλευτέ, αλλά όσοι είναι. Ο κ. Κόλμαν από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλου. Με την άδειά σα, Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχά στην συνάδελφο από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, που ήταν η επικεφαλή υπηρεσία τη διαπραγμάτευση, για να σα δώσω το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαπραγματευθήκαμε αυτή τη συμφωνία και συνεχεία θα πάμε στα ειδικά σημεία τη συμφωνία αυτή και θα σου κάνω ένα πρόβλημα, λέει πρόεδρος, όταν είσαστε λακωνικοί και οι δύο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Εγώ θα είμαι λακωνική. Ναι, καλωσορίζουμε την σύμφωνη γνώμη της ΑΦΕΤ προχθές και περιμένουμε να δώσετε κι εσείς τη σύμφωνη γνώμη σας. Και ελπίζουμε και η Ολομέλεια ε, πριν τελειώσει αυτή η κοινοβουλευτική θητεία. Όπως είπε και η συγκήτρια, όλα τα κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει πλέον την συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασίας. Θα τεθεί σε ισχύ λοιπόν αμέσως μετά την σύμφωνη γνώση του, γνώμη του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η Συμφωνία εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας δεν είναι Συμφωνία Επανεισδοχής αυτή καθ' αυτή. Έχει μια ρήτρα επανεισδοχής απλώς που ανοίγει τη δυνατότητα τα συμβαλόμενα μέρη να διαπραγματευτούν μια συμφωνία επανεισδοχής στο, στο μέλλον, αλλά δεν είναι η ίδια συμφωνία επανεισδοχής. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με την Ινδονησία είναι η πρώτη τέτοια συμφωνία με χώρα ε, της Νοτιοανατολικής Ασίας που περιλαμβάνει ρήτρα επανεισδοχής. Δίδουμε μεγάλη σημασία στην ε, Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία. Θέλουμε να μπει γρήγορα σε εφαρμογή, γιατί μα δίνει δυνατότητα για περισσότερη συνεργασία με την Ινδονησία και για θέματα μετανάστευσης βεβαίως και οι διμερείς μας σχέσεις νομίζω θα φτάσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο χάρη σε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ, ο κύριος Κόλμαν. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω πολύ σύντομα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της, μακρόπνοη. Υπάρχουν κάποιες γενικές συστάσεις που αφορούν ε, σε ευρύτερα θέματα πολιτικής επανεισδοχής Όπω είπε και συνάδελφό μου, είναι μια πολύ περιορισμένη ρήτρα επανεισδοχή και δεν μπορεί να συγκριθεί με μια πραγματική συμφωνία επανεισδοχή, όπου έχουμε ε, διατάξεις για τις διαδικασίες, τις προθεσμίες για να λάβει κανείς πίσω τους συμμεταπούς και τους απάτριδες. Σε αυτή τη ρήτρα ασχολούμαστε με την επανεισδοχή των ημεδαπών. οι συστάσει τη ηγήτρια είπε να λάβουμε υπόψη μα ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει μια συμφωνία 100% για την επανεισδοχή στο μέλλον. Την σημειώνουμε αυτή την σύσταση. Αλλά δεν υπάρχει σχέδιο από πλευρά Κομισιόν να κάνουμε κάτι τέτοιο για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχουν πολύ λίγοι παράτυποι μετανάστε από την ε, Ινδονησία, δηλαδή Ινδονήσοι που φτάνουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τη διέλευση, δεν έχουμε τα ακριβή στοιχεία, αλλά πιστεύουμε στοιχηματίζουμε ότι οι περισσότεροι παράτυποι μετανάστες που διέρχονται μέσω της Ινδονησίας και φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να φτάσουν να προχωρήσουν, να πάνε στην Αυστραλία ίσως. Ή μάλλον δεν πάνε οι περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στην Αυστραλία. Από την Ελληνική Προεδρία θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο για να σχολιάσει. Δεν έχω τα ονόματά σας εδώ. Όχι. Ο κύριος Μπρόνς. Μία γρήγορη ερώτηση. Λακωνικός θα είμαι. Καταλαβαίνω το πεδίο εφαρμογή της ε, Συμφωνίας Επανεισδοχής όταν μιλάμε για τρίτες χώρες. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται για τους ε, ημεδαπούς Υπάρχει καμία χώρα δηλαδή που αρνείται να πάρει πίσω τους μεταπούς της, τους πολίτες της. Να απαντήσει η συγγήτρια. Κυρία Γκόμες, θέλετε να απαντήσετε και να ολοκληρώσετε κιόλα με τα καταληκτικά σας σχόλια. Νομίζω ότι η ερώτηση είναι ότι η υπηκότητα θα πρέπει καταρχάς να μπορεί να ταυτοποιηθεί. Γιατί για πολλούς ανθρώπους που διέρχονται από την Ινδονησία, οι περισσότεροι δεν θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουν να πάνε στην Αυστραλία. Το είπε αυτό η Κομισιόν. Αλλά πολλοί από αυτούς είναι απάτριδες. Ή που είναι ασαφής η εθνικότητά τους. Καταληκτικά θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Γκόμες. Mm. Να τονίσω ότι χρειαζόμαστε μια πραγματική διαπραγμάτευση για να φτάσουμε σε μια πλήρη συμφωνία δοχής. Αλλά είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά έχουμε βάλει μια τέτοια ρήτρα σε συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να έχει κανένα δισταγμό το Κοινοβούλιο για να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Είναι κάτι που ανοίγει το δρόμο για μια πραγματική συμφωνία επανεισδοχή. σω σε αυτή τη φάση δεν έχουμε ανάγκη για μια τέτοια συμφωνία, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανεί. Εγώ είδα και έζησα εποχές όπου υπήρξαν τέτοιες κρίσει στην Ασία που επηρέασαν όχι μόνο τις ασιατικές χώρες, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό, μπορεί να γίνει σημαντικό στο μέλλον. Και μια και η Ινδονησία συμφωνεί, θα πρέπει να δώσουμε τη συμφωνή γνώμη μας. Ευχαριστώ. Προθεσμία για τροπολογίες είναι 30 Ιανουαρίου. Μόνο ε, διαδικαστικές τροπολογίες θα δεχτούμε και θα ψηφίσουμε 12-13 Φεβρουαρίου. Το επόμενο σημείο προβλέπετε να αρχίσετε στις 11. Έχουμε όμως τον κύριο Σόμερ που είναι ο ένας από τους εισηγητές. Ο κύριος Ένσιου δεν είναι ακόμα εδώ. Φοβάμαι ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 11. Okay. See you back at 11. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Αρχίζει η συνεδρίαση μετά την ολιγόλεπτη διακοπή. Παρακαλώ, αν θέλετε να συζητήσετε, κάντε το έξω. Επόμενο και τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα είναι μια κοινή συζήτηση για τα έξυπνα σύνορα. Το πακέτο λοιπόν των έξυπνων σύνορων αποτελείται από τρεις διαφορετικές εκθέσεις. Το πρόγραμμα καταχώρηση ταξιδιωτών με εισηγητή τον κύριο Ένσιου, το συστημα καταχώρηση καταχώρησης εισόδου-εξόδου με εισηγήτρια την κυρία Ζόμαρ και η κοινή έκθεση για την τροποποίηση του κανονισμού 562-2006 όσον αφορά την χρήση του συστήματος εισόδου-εξόδου και του προγράμματος καταχώρησης ταξιδιωτών. Η τελευταία συζήτηση για το πακέτο των έξυπνων συνόρων έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι συγκεκριτές παρουσίασαν τα έγγραφα εργασίας τους. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων και ως συνέχεια αυτή θα ήθελα να καλέσω τους εισηγητές να λάβουν το λόγο. Ποιο θέλει να αρχίσει, η κυρία Ένσιου ή η κυρία Σόμερ. Κυρία Ένσιου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε τους τελευταίους πέντε μήνες από την πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή Λίμπε για το πακέτο των έξυπνων συνόρων αφιερωθήκαμε σε τεχνικού ύφους συζητήσεις. Και κάναμε και δύο επιτόπιες επισκέψεις στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και στα ρωσικά σύνορα. Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα από αυτές τις επισκέψεις και βοήθησαν τη δουλειά των εισηγητών. Επίσης, φάνηκε ότι έχουμε ορισμένα προβλήματα θεμελιωδών ζητημάτων με την πρόταση της Επιτροπής. Επίσης χρειάζεται περιττέρω διευκρίνηση ορισμένων στοιχείων. Θεωρώ ότι η αναλογικότητα και η προστιθέμενη αξία που αναμένεται και για το σύστημα εισόδου-εξόδου και για το σύστημα καταχώρησης ταξιδιωτών, έτσι όπως είναι σήμερα, δεν έχουν φανεί επαρκώς. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της εσύστασης αυτής και με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου να διεξάγει μια μελέτη η οποία θα εξετάσει ε, την εφικτότητα των δύο αυτών προτάσεων, το, την εφικτότητα του κόστους και την, ε, το πόσο υλοποιήσιμες είναι. Ωστόσο πιστεύω ότι η μελέτη αυτή θα επιτύχει το στόχο της μόνο όταν οι δύο συνομοθέτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνήσουν για το πεδίο εφαρμογή όσον αφορά τα σημεία αναφοράς. Επομένως, θεωρούμε ακατάλληλο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατάλληλο. Ακατάλληλο μάλλον τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι μόνο παρατηρητές τη όλη διαδικασία, έτσι όπω έχει αναφέρει πολλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη, γι' αυτό και θα έπρεπε να είναι πλήρω εντάμενο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη συζήτηση για τα επόμενα βήματα σχετικά με, τις, ε, το μέλλον των τριών αυτών εκθέσεων. Τα μέτρα που προτείνονται και θα έχουν ενδεχομένως ε, εκτεταμένες συνέπειες και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται πλήρως στην απόφαση και οι δύο συνομοθέτες. Να τονίσω επίσης ότι είναι παράδεκτο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να οργανώσει εργαστήριο για τον ορισμό του πεδίου εφαρμογή της μελέτης αυτής μια Παρασκευή, την Παρασκευή στις 5 Φεβρουαρίου, την 7 Φεβρουαρίου, διορθώνει ο συγητής, την επόμενη της τελευταίας ημέρας ολομέλειας του Στρασβούργου. Αυτό το κάνει αδύνατο για τους περισσότερους ευρωβουλευτές να παρευρεθούν στο εργαστήριο αυτό. Οι εισηγητέ, λοιπόν και οι εισηγητέ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωση μιας κοινή προσέγγισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους στόχους και το πεδίο εφαρμογή της μελέτης και του πιλωτικού προγράμματος και θεωρούμε ότι ως συνομοθέτες η άποψή μας και οι προτάσεις μας πρέπει να συμπεριληφθούν πλήρως στην επερχόμενη διαδικασία. Και όλο το project πρέπει να εστιάσει σε ορισμένα βασικά θεμελιώδη ζητήματα της πρότασης, όπως το χρονοδιάγραμμα για τα δύο συστήματα. Το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα λοιπόν πρέπει να επανεξεταστεί, ιδιαίτερα και το σύστημα εισόδου-εξόδου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ε, όλα τα διάφορα σενάρια που θα εξεταστούν. Επίσης, η μελέτη εφικτότητας που θα εξετάσει τη δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν το σύστημα εισόδου-εξόδου και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν τα κράτη-μέλη και αν τον διαθέτουν. Επίσης, η μελέτη πρέπει να εξετάσει το πόσο είναι εφικτή αυτή η έλεγχη βιομετρικών δεδομένων στα χερσαία και θαλάσσια και αέρια σύνορα, ιδιαίτερα όσον αφορά τους χρόνους αναμονής και επεξεργασίας των δεδομένων των επιβατών αυτών. Η μελέτη αυτή, επίσης, θα πρέπει να εξετάσει αν το σύστημα ΒΙΣ, το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, έχει τη δυνατότητα να ε, συμπεριλάβει μια λειτουργία εισόδου-εξόδου που θα συμμορφώνεται με την οδηγία και την προστασία των δεδομένων των επιβατών. Επίσης, χρειάζεται να γίνει μια νέα ανάλυση κόστους. Το εκτιμόμενο κόστος και για το σύστημα καταχώρηση εξοδου, ε, εισόδου και για το πρόγραμμα καταχώρηση ταξιδιωτών υπολογίστηκε με ένα ποσοστό λάθος 25%. Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι οικονομικοί περιορισμοί στις μετά από τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης η μελέτη πρέπει να παρέχει μια εκτίμηση αντικτύπου για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ε, χρήση των βιομετρικών δεδομένων των επιβατών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης πρέπει να διαβεβαιώσει το ε, Κοινοβούλιο ότι η συμμετοχή του θα εγγυάται και, θα... και δεν θα παραλυφθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζόμερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον ε, κύριο Έντσιου. Να πω ότι η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ, με τη σειρά μου, θα ήθελα να, να τονίσω ότι μετά από τις τελευταίες συνομιλίες στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχουν γίνει πάρα πολλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ακούσατε τίποτα εμείς δεν κάναμε και τίποτα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Να σας υπενθυμίσω ότι περίπου το 90% των μελών αυτής της Επιτροπής διάβασαν το σχέδιο πρότασης και δεν έμειναν ευχαριστημένοι. Και αυτό λοιπόν ήταν η αφορμή για να επανεξετάσουμε το θέμα με μεγάλη προσοχή. Χαίρομαι πολύ που έχουμε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος από το Συμβούλιο. Είναι κάποιος. Ακόμα καλύτερα. Θαυμάσια. Μπορούμε λοιπόν να ακούσουμε και την άποψη και των δύο πλευρών. Είναι λοιπόν ένα πολύ περίπλοκο και τεχνικό θέμα το πακέτο για τα έξυπνα σύνορα. Είναι λοιπόν σημαντικό να αποκτήσουμε μια εικόνα του τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι πρακτικές. Και ο συνάδελφος Ένσιου ήδη σας έκανε την εισήγησή του. Ήδη σας παρουσίασε λοιπόν τα... το τι έγινε. Ήμασταν στο Άμστερνταμ Είδαμε τη λειτουργία των e-gates, των ηλεκτρονικών πυλών, είδαμε την πιλωτική εφαρμογή λοιπόν του προγράμματος καταχώρησης των ταξιδιωτών και αποκομίσαμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εικόνες. Μπορέσαμε λοιπόν να αποκτήσουμε μια εικόνα του τι περίπου γίνεται και πώς εφαρμόζεται στην πράξη ο συνοριακός έλεγχος. Και λίγο πριν τα Χριστούγεννα πέρυσι Πήγαμε στη Φιλανδία, στα ρωσικά σύνορα. Και διότι κατέστησα σαφέ ότι δεν έχει νόημα να κοιτάζουμε μόνο τα αεροδρόμια, πρέπει να δούμε και τι γίνεται στα χερσαία σύνορα. Πήγαμε λοιπόν εκεί και πραγματικά είδαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό κίνησης ταξιδιωτών ανάμεσα στη Φιλανδία και τη Ρωσία μου μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία που αποκομίσαμε, διότι είχαμε την εντύπωση ότι τα σύνορα είναι απομονωμένα. Καμία σχέση όμως τα σύνορα αυτά διασχίζονται από πολλού ταξιδιώτε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο συνοριακό έλεγχος να γίνεται γρήγορα έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και μεγάλες ουρές. Επίσης εκεί στη Φιλανδία κέντρο... Κεντρικό αντικείμενο ήταν το σύστημα καταχώρησης εισόδου-εξόδου. Μελετήσαμε λοιπόν το σύστημα αυτό και αυτή τη στιγμή συντάσσουμε την έκθεση σχετικά με τις εμπειρίες μας στη Φιλανδία και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, Φιλανδούς ε, συναδέλφους οι οποίοι μας βοήθησαν στην ε, μελέτη μας. Είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις προς τους συνοριοφύλακες και μας απάντησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. <coughs> Λάβαμε λοιπόν πάρα πολλές πολύτιμες, εξαιρετικά πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες μας βοήθησαν στην δουλειά μας εδώ, στη δημιουργία των εκθέσεων. Πριν ε, πάμε όμως στη Φιλανδία συναντηθήκαμε με εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους κοιόδης εισηγητές. Έγινε λοιπόν αυτή η πρόταση έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται με τη μελέτη και με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πολύ θετική αντίδραση είχε παρακολουθήσει και όλα στη συζήτηση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και αποφασίστηκε μετά από την ε, μελέτη αυτή να εφαρμοστεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε κάποιο κράτος μέλος. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας ενημερώσει για αυτό περαιτέρω. Όσον αφορά τώρα την τεχνική εφαρμογή του συστήματος, υπάρχουν διάφορα που χρειάζεται να διευκρινιστούν. Καταρχάς πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, εάν χρειάζεται ένα εντελώς νέο σύστημα με εντελώς νέο τρόπο συλλογής δεδομένων ή αν μπορούμε να βελτιώσουμε το υπάρχον σύστημα. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία θα εξετάσει η μελέτη που θα γίνει και ελπίζω, όπως είπε και ο συνάδελφος Ένσιου, να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο ρόλος μας ως συνομοθέτη. Και όπως είπε και ο συνάδελφος κύριος Ένσιου, η 7η Φεβρουαρίου είναι μια ατυχής ημερομηνία. Είναι μια μέρα μετά την τελευταία μέρα ολομέλειας του Στρασβούργου και δεν μπορούμε να είμαστε λοιπόν στις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν μας είπε ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ήταν η μοναδική ημερομηνία που μπορούσε να γίνει αυτό το εργαστήριο. Όμως, εγώ θα ήθελα εδώ να αντιπροτείνω να γίνει μια πρώτερη συνάντηση, έτσι ώστε να συζητήσουμε για αυτό το εργαστήριο, για το τι θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου, να μας ενημερώσουν. Τώρα από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η μελέτη δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν και αμέσως να εφαρμοστούν αποφάσεις για τα έξυπνα σύνορα. Εμείς αυτό που επιθυμούμε είναι να μην γίνουν βιαστικές ενέργειες αλλά να υπάρξει ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα για τον συνοριακό έλεγχο. Ήδη ο συνάδελφος ανέφερε και τα προβλήματα που θα μας απασχολήσουν, που μας έχουν ήδη απασχολήσει από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι εδώ. Το πακέτο για τα έξυπνα σύνορα δεν πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν, τότε πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και κατέστη σαφέ μετά από την επίσκεψή μας στη Φιλανδία ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικούς συνοριακούς ελέγχους και ένα διαφορετικό σύστημα. Το σύστημα των ε, σφραγίδων στα διαβατήρια, στα ταξιδιωτικά έγγραφα των επιβατών είναι πεπαλαιωμένο. Γι' αυτό χρειάζεται ένας εξυγχρονισμός που να συμμορφώνεται με τα σύγχρονα, τα νεότερα τεχνικά πρότυπα. Είναι πραγματικά, ε, είναι πραγματικά το πόσοι ταξιδιώτες διασχίζουν αυτά τα σύνορα Φιλανδίας-Ρωσίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να ε, διεξάγουμε τους συνοριακούς ελέγχους ε, το ταχύτερο δυνατόν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ίσως συμπεριληφθούν τα βιομετρικά δεδομένα, τα δακτυλικά αποτυπώματα ή τα σκάν ε, της σύριδας του ματιού. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν αυτά μπορούν να ληφθούν υπόψη, να μπορούν να συμπεριληφθούν το πόσο είναι εφικτά και από πλευράς χρόνου και από πλευράς τεχνολογίας και κόστους. Από την άλλη, στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και ιδέες για ένα νέο σύστημα ε, ελέγχων με την χρήση νέων τεχνολογιών το οποίο μπορούμε να δούμε ή αν μπορούμε να το συνδυάσουμε με το υπάρχον σύστημα ή αν μπορούμε να κοιτάξουμε περισσότερο προς το μέλλον και δημιουργήσουμε κάτι καλό, κάτι που να έχει λάβει υπόψη του όλε τις τεχνικές εξελίξεις, διότι το τελευταίο που θέλουμε είναι όταν επιτέλους εφαρμοστεί αυτό το σύστημα να έχει ήδη παλιώσει. Πρέπει επομένως πραγματικά να είμαστε ενήμεροι για τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, Υπάρχουν στο μεταξύ 13 ε, χώρες ε, του χώρου του Σέγγεν που έχουν ένα δικό τους ε, σύστημα καταχώρησης εισόδου-εξόδου ταξιδιωτών. Πρέπει να δούμε αν μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα συστήματα. Στη Φιλανδία είδαμε ότι το σύστημα αυτό που χρησιμοποιούν λειτουργεί πάρα πολύ καλά και όμως αυτό που λείπει από το σύστημα είναι το πού πηγαίνει ο ταξιδιώτη μετά τη Φιλανδία, αφού φύγει από τη Φιλανδία. Γι' αυτό λοιπόν το νέο σύστημα που θα δημιουργηθεί πρέπει να μας επιτρέπει να βλέπουμε το δρομολόγιο των ε, ταξιδιωτών, όχι μόνο το σημείο εισόδου και το πού πηγαίνουν εντό της επικράτειας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σα είπα, 13 χώρες έχουν ήδη ένα δικό του σύστημα καταγραφής εισόδου-εξόδου. Έχουν διαφορετικές ε, τεχνικές ε, λεπτομέρειες ε, τα συστήματα αυτά και θα μπορούσαμε ίσως να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συνδυαστούν αυτά τα συστήματα και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ή από την αρχή ή με συνδυασμό των ήδη υφισταμένων συστήματων που χρησιμοποιούν αυτά τα κρατημέλη. Και αν δεν κάνω λάθος, πριν από πολλά χρόνια υπήρξε και μία έκθεση για τις τεχνικές προδιαγραφές και την διαλειτουργικότητα των τεχνικών συστημάτων τα οποία έχουν ε, δημιουργηθεί χωρίς ε, πρώτα να συνδέονται το ένα με το άλλο. Ανεξάρτητα λοιπόν συστήματα και το πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε. Υπήρξε μια τέτοια έκθεση πριν από κάποια χρόνια στο Κοινοβούλιο. Τώρα, στο μεταξύ, όλες μας οι εμπειρίες, όλες μας οι συζητήσεις για το θέμα αυτό δείχνουν ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα σύστημα καταχώρησης εισόδου-εξόδου, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πραγματικά με τις σφραγίδες εισόδου και εξόδου. Αυτό είναι χρονοβόρο και ε, προβληματικό σύστημα, απαιτεί πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς πρέπει να δούμε πώς ε, αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο. Όπως είπε και ο συνάδελφος Έντσι, χρειαζόμαστε νέα εκτίμηση κόστους. Δεν μας φαίνεται ρεαλιστικός αυτός ο υπολογισμός που έχει ήδη γίνει. Και φυσικά υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν και την ε, δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα εφαρμογής αυτών των ε, πιλωτικών προγραμμάτων και να μην ξεχνάμε ότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, είναι υψή της σημασίας και πρέπει οπωσδήποτε να είναι το κύριο μέλημά μας το πακέτο για τα έξυπνα σύνορα. Όλα αυτά φυσικά όλες αυτές τις προτάσεις και τις επιθυμίες μας θα τις ε, γνωστοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τους ε, στείλουμε έναν λεπτομερή κατάλογο τον οποίο ελπίζω να συμπεριλάβουν υπόψη ε, μετά στα αποτελέσματα της μελέτης τους για το πακέτο των έξυπνων συνόρων και ελπίζω να καταφέρουμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες πριν τις 7 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου να σχολιάσουν σύντομα ε, το θέμα αυτό, ιδιαίτερα την ημερομηνία που έχει προταθεί, την 7η Φεβρουαρίου. Προτείνω η, Επιτροπή, η Γραμματεία της Επιτροπής να στείλει το ε, χρονοδιάγραμμα των ε, συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή. Εντάξει, λάθη μπορούν να γίνουν, όμως ελπίζω να σταματήσουν να γίνονται στο μέλλον. Κύριε Πόου, εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Λέγω Φρανκ ε, Πό, είμαι τμήματάρχη των, των διευρωπαϊκών ε, συστημάτων και την ε, σχέση του με το Γιουλίσα. Είμαι επικεφαλής της Task Force της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών για την παράτυπη μετανάστευση και Είμαι υπεύθυνη για το Eurodac, το VIS, το VIS και το SIS2. Γνωρίζω πάρα, πολύ, πάρα πολλά πράγματα για το εγχείρημα όπως αυτό και με πολύ σεβασμό και ταπεινοφροσύνη αντιμετωπίζω το στόχο μας. Διδαχθήκαμε πικρά μαθήματα από την ανάπτυξη των συστημάτων και τα μαθήματα αυτά τα πικρά θα λυθούν σίγουρα υπόψη. Μετά από αυτά, η Κομισιόν φυσικά εκτιμάει πολύ την υψηλή σημασία που δίνει το Κοινοβούλιο στο πακέτο αυτό. Πολύ σύντομο μπορούμε, μπορώ να είμαι. Από όλα όσα άκουσα από την εισηγήτρια και τον, τους δύο εισηγητές μάλλον, ε, δεν βρίσκω παράλογο, δεν διαφωνώ μαζί του και η πρόθεσή μας όντως είναι να λάβουμε υπόψη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις προτάσεις και υποδείξεις που έγιναν για τη μελέτη αυτή. Με την επιφύλαξη των θεσμικών προνομίων της Κομισιόν, θέλω να σας πω ότι θέλουμε και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις απόψεις των συνομοθετών 100% εάν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς και να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Και φυσικά το θέλουμε, γιατί είμαστε όντως πεπισμένοι για τους λόγους που ανέφερε η κυρία Σόμε, ότι είναι απολύτως αναγκαίο να προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε στο μέλλον τη διαχείριση των συνόρων μας. Γίνεται ατυχής, η χρήση, ατυχής χρήση της λέξης ε, παρατηρητής. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο όπως συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε, Πρόεδρε, για την επιλογή το, της ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου, που δεν ήταν καλή επιλογή. Δεν θα ξανασυμβεί. Προσφερθήκαμε να συναντηθούμε όμως με τους εισηγητές, όσες φορές χρειαστεί. Πριν από τη συνάντηση, για να λάβουμε υπόψη της απόψας. Θα υπάρξει και βοήθεια. Η συνάντηση, από ό,τι ξέρω, θα είναι μια τεχνική φύσεως συνάντηση, δεν έχει νόημα τώρα να μιλήσουμε για αυτή τη φάση για πολιτικές επιλογές, οι οποίες θα γίνουν αργότερα, λαμβάνοντας υπόψη τους ρόλους των θεσμικών οργάνων. Δεν πρέπει να είναι η εκδήλωση της χρονιάς αυτή ούτως ή άλλως. Και δεν θα γίνει τίποτα άλλο μετά. Όχι. Θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις και άλλες χρονικές στιγμές όπου θα μπορέσετε να μας μιλήσετε για το περιεχόμενο της μελέτης και ελπίζουμε όταν να ξεκαθαριστεί περισσότερο το πεδίο της ε, έκθεσης θα λάβουμε υπόψη μας απόψη και των δύο συνομοθετών και των υπολείπων. Μου είπατε να είμαι λακωνικό. Δεν, αρκούν, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερα. Επί τη ουσία σας είπα ότι συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν. Να τονίσω ειδικά δύο πράγματα. Το κόστο, πρέπει να το λάβουμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το διαφορετικό πλαίσιο στο οποίο ε, κινούμαστε σήμερα και η οικονομική κατάσταση είναι διαφορετική και ο προπολογισμό διαφορετικό. Και στο μεταξύ επίση μην πω ότι κάθε μήνα γίνονται νέε εξελίξει στα κράτη-μέλη. Νέε αυτοματοποιημένε πύλε που δείχνουν και την πίεση που υπάρχει στα σύνορα, γιατί αλλιώ τα κράτη-μέλη θα προβαίνουν σε τέτοιε επιλογέ. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε γίνεται ξαναχρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σε οποιαδήποτε μελλοντική τεχνική συσκευή που αναπτύσσεται. Ευχαριστώ, κύριε Πολ. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας συγχαρώ για τα νέα σας καθήκοντα ή να σας ευχηθώ α, καλή δύναμη. Από μέρους της Ελληνικής Προεδρίας. Παρακαλώ. Yes, good morning, Mr. President, thank Καλημέρα και ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Μια και υπάρχει ελληνική διερμηνία, θα ήθελα να μιλήσω στη μετρική μου γλώσσα, παρακαλώ, μου επιτρέπετε θα σας δώσω μία γενική επισκόπηση των ε, τρεχουσών εργασιών στο Συμβούλιο, πολύ σύντομα και πολύ λακωνικά, ε, λέγοντας ότι ως γνωστόν αυτοί, αυτές οι νομοθετικές προτάσεις έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή τον ε, περασμένο Μάρτιο. Έκτοτε συζητιούνται αναλυτικά και σε βάθος στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στην ομάδα εργασίας για τα σύνορα και η Προεδρία έχει ήδη ξεκινήσει άτυπες επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο αυτών των προτάσεων. Από την έναρξη της Προεδρίας μας έχουν γίνει δύο συνεδριάσεις σε επίπεδο συμβούλων δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και οι συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί στην ανέβρεση του κατάλληλου τρόπου, της κατάλληλης προσέγγισης για να προχωρήσουμε εμπρός στις εργασίες των νομοθετικών αυτών προτάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η Προεδρία έχει συντάξει και έχει θέσει προς διαβούλευση και συζήτηση ένα δικό της σχέδιο α, προσέγγισης, το οποίο βασίζεται στη γνωστή σε όλους σας πρόταση της Επιτροπής, έχοντας συμπεριλάβει και παρατηρήσεις και σχόλια των κρατών μελών. Η πρόθεσή μας είναι αυτή η προσέγγιση να συζητηθεί, να τύχει αποδοχής και να πάει στο κορεπέρ για πολιτική υιοθέτηση. Νομίζω αυτό δίνει το στίγμα των εργασιών του Συμβουλίου και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να πω ότι βεβαίως όλα όσα υπόθηκαν, με όλα όσα υπόθηκαν είμαστε και εμείς σύμφωνοι. Κανείς δεν παραγνωρίζει φυσικά το ρόλο του συνομοθέτη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξυπακούεται ότι πρέπει να έχει λόγο και ρόλο και βεβαίως νομίζω ο σκοπός όλων είναι κοινό και η στόχευση κοινή ε, για την επιτυχία των νομοθετικών εγχειρημάτων και την ευόδοσή τους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε. Τρεις ευρωβουλευτές ζητούν το λόγο και εγώ. Ο κ. Κοέλιο επίσης. Ποιος άλλος? Ο κ. Κέρκο. Τέσσερις ομιλητές. Ο κύριος Κέρκχοπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα-δύο σημεία θα ήθελα να θίξω. Ενώ υποστηρίζω εν γέννη απόλυτα αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία, θέλω να είμαι σίγουρος, γιατί άκουσα την κυρία Σόμερ για τις επισκέψεις κτλ. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι έχουμε επωφεληθεί όσο μπορούσαμε από τις εμπειρίες που είχαν άλλοι, ε, ειδικά με τα έξυπνα σύνορα. Ειδικά τα έξυπνα σύνορα μεταξύ ε, Αμερικής και Καναδά, Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, όπου υπάρχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά με αυτά που προτείνουμε εδώ. Νομίζω ότι εν γέννη η προσέγγιση είναι επιτυχής. Αλλά έχω μία ανησυχία για την τεχνολογία σήμερα και τη χρήση της. Και σε ποιο βαθμό οι αποτυχίες στη νέα τεχνολογία, που είναι πασίγνωστες σε όλες τις χώρες μας και στα θεσμικά όργανα, αποτυχίες τρομακτικές που κόστησαν εκατομμύρια, όπου η μοναδική τυχερία που υποφελήθηκαν ήταν η εταιρεία software. Θέλω να είμαι σίγουρος 100% ότι δεν πρόκειται να επιλέξω μια γελία λύση όπου θα ξοδέψουμε απίστευτα λεφτά, θα κάνουμε τρομακτικά λάθη. Ξέρω ότι έχουμε όλα αυτά, όλη αυτή η χαρτούρα ε, για το σύστημα εισόδου-εξόδου και τα κτλ. Και γελιοποιούμε, ας πούμε, τα, το υπόθεμα χάρτου και πάντα θεωρούμε ότι «Oh, wow, τα κομπιούτερ είναι καλύτερα». Αλλά Καμιά φορά κάνουμε τρομακτικά λάθη με το κομπιούτερ και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να διορθώσει. Αυτό έγινε στο χρηματοπιστωτικό τομέα, σε διάφορους τομείς, όπου και να σκεφτώ έχει γίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, τι θέλω να πω. Έχουμε ε, λάβει υπόψη μας την εμπειρία άλλων που έχουν προχωρήσει σε αυτόν τον τομέα, όχι μόνο τη δική μας. Και θα εξασφαλίσουμε με συνετό τρόπο τη χρήση της τεχνολογίας και δεν θα καταλήξουμε να γελιοποιούμαστε ακόμα, να γελιοποιηθούμε ακόμα μια φορά όπως γελιοποιηθήκαμε στο παρελθόν. Μου άρεσε η αναλυσή σας, κυρία Κέλλερ. ενδιαφέρον που λέει το Συμβούλιο και, και η Κομισιόν. Είσαστε τόσο σημαντικοί, θα σας λάβουμε υπόψη κτλ. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει θα σας λάβουμε υπόψη στο βαθμό του δυνατού. Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συμφωνήσαμε να καθυστερήσουμε αυτή την νομοθετική διαδικασία. Υπό... Μέχρι να έχουμε τη μελέτη που θα λάβουμε υπόψη ε, και θα μας λάβετε υπόψη σας ε, ισοτιμία με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Αν θέλετε λοιπόν πιο θετική στάση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μας λάβετε υπόψη σας στα σοβαρά. Ε, το, είχαν, ε, το είχε προτείνει και ο προκάτοχός σας κύριε Μπορατίνη, αν το προφέρω σωστά το όνομά του. Ε, μας, απο, μας αποκαλείτε παρατηρητές, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει τίποτα. Θέλουμε ίση μεταχείριση η, Κομισι... η Κομισιόν θέλει στενή συνεργασία με το Συμβούλιο, αλλά όχι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί είμαστε εδώ πέρα και ακούμε απλώ από άλλου, α πούμε, ότι έχουν γίνει πολλέ συναντήσει μεταξύ Κομισιόν και Συμβουλίου. Ο κ. Μπορατίνσκι μα είπε ότι η Κομισιόν θα στι 15 με 16 ε, Ιανουαρίου θα στείλει ένα κείμενο με την μελέτη και θα τη στείλει στο Συμβούλιο και σε εμάς. Τα κράτη-μέλη λάβανε αυτό το έγγραφο, αλλά όχι εμεί. Σα παρακαλώ, διορθώστε το λάθο στο το συντομότερο δυνατόν. Επίση, η Κομισιόν δεν μα προσκάλεσε στην πρώτη συνάντηση για να συλλέξει στοιχεία για, το, για τη μελέτη. Δεν νομίζω ότι θα είναι και τόσο τεχνικό αυτό το, αυτή τη συνάντηση. Θα καθορίσει το πεδίο της ε, μελέτη. Είναι πολύ σημαντικό και το πιλωτικό σχέδιο θα αποτελέσει σταθμό για να δούμε Πώ θα προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα. Αυτή η συνάντηση δεν είναι τεχνική, αλλά θα καθορίσει το πεδίο της μελέτης. Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι πότε δεν μπορούμε να έρθουμε και εσεί πότε την κανονίσατε Παρασκευή Στρασβούργου. Κανονικά θα πρέπει να την ακυρώσετε και να την βάλετε μια άλλη ημερομηνία. Και αν το κάνετε, ε, προσέξτε να μην αφήσετε και εντελώ κατά τύχη έξω το σκιώδη ηγητή των πρασίνων. Ε, να μας προσκαλέσετε και εμά, παρακαλώ εκεί. Ποιο είναι το πρόβλημα μια στιγμή γιατί υπάρχει κι άλλο, είμαι σίγουρη. Σας στείλαμε επίσης ε, ένα κατάλογο, όχι επιθυμιών, αλλά κάτι για το οποίο είναι εκ των όνων κάνευτο κοινοβούλιο. Ε, είναι η πρόταση που να λαμβάνει υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα τα Και, και να μην ε, λαμβάνει υπόψη μόνο μία λύση, αλλά διάφορες λύσεις, όχι μόνο τεχνολογικές. Όλες αυτές οι επιλογές θα πρέπει να διερευνηθούν και θα ήθελα να ακούσω περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς λαμβάνεται υπόψη αυτές τις ε, πολύ συγκεκριμένες απαιτήσει ε, του Κοινοβουλίου υπόψη. Για μας ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό να μην κουνηθούμε ούτε ένα γιώτα από αυτή τη στάση, από αυτή τη γραμμή. Αυτά που μας είπε η συγκίτη είναι πολύ σημαντικό, σημαντικά. Αλλά αν δεν απαντήσει στα όσα ζητάμε η Κομισιόν, θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αυστηροί, να πάμε το θέμα στους συντονιστές, να είμαστε πιο απαιτητικοί κτλ. Και ελπίζω να με υποστηρίξουν οι ε, συναδελφοί μου ε, προς αυτήν την κατεύθυνση. Εάν δεν δεχτεί η Κομισιόν τα αιτήματά μας. Σας συγχαίρω βέβαια για την νέα σας θέση, ε, πρόσωπε της Κομισιόν. Ε, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να βρείτε τον μπούσουλα τις πρώτες σας μέρες, τη νέα σας θέση, αλλά ελπίζω, όσο δύσκολο και αν είναι, να ανταποκριθείτε στα αιτήματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκοέγιο. Thank you ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω την μελέτη. Όπως είπε η κυρία Κέλλερ, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες και ελπίζουμε ότι τώρα θα μπορέσει το Κοινοβούλιο με δεδομένη αυτή τη μελέτη να λάβει κάποιες αποφάσεις. Όπως είπε ο κύριος Φρανκ Πομ. Οπότε και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αντλήσει κάποια διδάγματα όπως έγινε στο παρελθόν και νομίζω ότι θα είναι αυτό το κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Και εγώ διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. για την αναγκαιότητα του συστήματος και η κυρία Σόμερ επίσης μας ανέφερε ότι αυτή η μελέτη δεν είναι πραγματικά μελέτη που θα οδηγήσει το Κοινοβούλιο σε ένα ναι ή σε ένα όχι θα πρέπει αυτή η μελέτη να μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα προβλήματα. Και έχουμε τέσσερα ζητήματα ε, στα οποία πρέπει να βοηθήσει αυτή η μελέτη. Πρώτα-πρώτα, Αυτέ οι εξαρχίες δεν είναι σαφέ το που θέλουμε να καταλήξουμε με αυτή τη δέσμη μέτρων. Μπορέσουμε τελικά να καταλάβουμε ποια είναι η προσθεμένη αξία του συστήματος. Δεύτερον, το κόστος. Όταν λέω κόστο, εννοώ το πραγματικό κόστο. Τα πρώτα αριθμητικά στοιχεία. Τα ξέρουμε, είναι εντυπωσιακά. Απρέπει να λάβουμε υπόψη τι γίνεται με το SIS2 γιατί ποτέ τα πρώτα στοιχεία δεν είναι τα οριστικά. Επομένως, αυτό θα πρέπει να κάνουμε με την μελέτη να προβλέψουμε πέραν των αρχικών δεδομένων να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος να έχουμε τέτοιο κόστος ως οριστικό κόστος του διαβήματος. κυρία Σόμερ μας μίλησε για την νέα τεχνολογία που ανοίγει πόρτες αλλά δημιουργεί κινδύνους. Για αυτό το θέμα η προστασία των ε, δεδομένων δεν μπορεί να είναι ένα θέμα που να θεωρείται δευτερεύον, είναι πρωτεύον και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Επίσης, σχέση μεταξύ των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, κρατών μελών. τι θα πρέπει να είναι η αρμοδιότητα της Ένωσης και τι θα είναι κάτι το οποίο θα αφορά τις εθνικές βάσεις δεδομένων. θα πρέπει να μας βοηθήσει αυτή η μελέτη σε αυτά τα τέσσερα ζητήματα. Να δούμε τι πάει καλά ή τι δεν πάει καλά. Που ολοχεύουν κίνδυνοι και που όχι. Επομένως, μια που έχουμε όλες αυτές τις επιφυλάξεις, ε, ό,τι πληροφορίες πάρουμε θα είναι χρήσιμες. Ευχαριστούμε εμείς, λέει η Πρόεδρος, και τώρα ο στον κατάλογο είμαι εγώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Πιστεύω ότι αυτή η μελέτη πρόκειται να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ακόμα εκρεμεί για μένα το θέμα του αν θα πούμε ναι, θα πούμε όχι. Αν ξεκινήσουμε όμως αυτή τη διαδρομή, τουλάχιστον να μπορέσουμε να την κάνουμε με τα λόγω γνώσεως. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ συμμερίζομαι τις αμφιβολίες του κύριου Κερχόβιτς. Φυλάξτε το. Γιατί ε, ακόμα δεν έχω δει κανένα μεγάλο πρόγραμμα που να το έχει πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά την πληροφορική και να είναι και σε κάποια πλαίσια προπολογισμού. Θα πρέπει να κλείσουμε επομένω συμπράσματα και από αλλού και από το παρελθόν. Γιατί έχουμε κάποια συστήματα παρόμοια που ήδη υπάρχουν. Είπατε το, θέμα, το, το, το σύστημα το αμερικανικό, το κρατικό. Από όσο γνωρίζω, κανένα από αυτά τα συστήματα δεν αποδίδει 100%. Ιδίω το αμερικανικό έχει παρουσιάσει πάρα πολλά προβλήματα. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Να προστατεύσουμε ας πούμε, το, κοινοβούλιο από ένα hacker που απλώς έχει στη διάθεσή του ένα φορητό υπολογιστή, λάπτοπ. Ναι, να, να αναθέσετε τα κριτήρια για τη μελέτη, αλλά σκεφτείτε πώς θα αποφύγουμε τις παγίδες στις οποίες πέσανε οι Αμερικανοί. Επίσης, για τα πιλωτικά προγράμματα. Δεν μου είναι τόσο σαφές το τι εννοούμε πιλωτικά προγράμματα. Ήδη τρέχει ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα στα Ακαδημία δεν μου αρέσουν καθόλου γιατί έτσι αυτοί με, με κοινωτικά χρήματα κάνουν αυτή τη δουλειά και έτσι δημιουργούν τελεσμένο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Επίσης νομίζω ότι ο πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπε ότι υπάρχει πίεση στα σύνορα και γι' αυτό το λόγο κάποιες χώρες θέλουν το σύστημα. Έτσι υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι. που μιλούμε για τόσο μεγάλη δαπάνη. Επισήμως θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει ποιος θα ωφεληθεί, ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν, ποιοι θα πάσουν αυτές τις υπηρεσίες, με ποιες εταιρείε έχετε συνομιλήσει ως Επιτροπή, ποιους λομπίστες. Δηλαδή, όχι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι και η αμυντική βιομηχανία που έχει σχέση και με τους Αμερικανούς οι οποίοι μας προμηθεύουν το σύστημα. Άρα αυτός ο οποίος το φτιάχνει, αυτός ο οποίος πρόκειται να τρέξει το σύστημα να δούμε τι, θα, θα σχετίζεται ε, θα, θα είναι στην Αμερική πού θα είναι. Αν δεν θέλετε να μας απαντήσετε εδώ και τώρα, τότε να κάνω επίσημο διάβημα. Συζητήσατε με κάποιες ε, εταιρείε. Ε, δεν είναι και τόσες πολλές. Σε όλο τον κόσμο λίγες είναι οι εταιρείε που φτιάχνουν τέτοια συστήματα τέτοιων διαστάσεων. Και δεν έχω μία εικόνα του τοπίου των οικονομικών συμφερόντων. Και του πού είναι εγκατεστημένες, που έχουν την έδρα τους οι σχετικές εταιρείες. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Να απαντήσω. Πρώτα απ' στον κύριο Κέρκοπ ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλα συστήματα αλλού στον κόσμο που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Είπα φέρετε το, το Αμερικανο-Καναδικά σύνορα. Έχω πάει και εκεί, έχω πάει και αλλού, σε άλλα σύνορα που χρησιμοποιούν παρόμοια συστήματα. Όμως είναι δύσκολο να συγκρίνουμε την κατάσταση που επικρατεί εκεί με την εδώ. Μια που Βγαίνει από τον Καναδά και μπαίνει στη ΣΥΠΑ. Οπότε το μόνο που χρειάζεται να κάνουν αυτές τις χώρες είναι να ανταλλάσσουν τα δεδομένα και αυτό και κάνουν. Και έχουν ένα σύμφωνο σχετικό το οποίο συνήφθη πέρσι. Καταλαβαίνετε ότι για μας δεν είναι τόσο καλή ιδέα να ανταλλάσσουμε δεδομένα με ας πούμε την Λευκορωσία όσον αφορά την είσοδο και έξοδο Όταν συμφωνείτε με αυτό, άρα επομένως δεν είναι συγκρίσιμες καταστάσεις. Και γι' αυτό και εξετάζουμε προσεκτικά τα συστήματα. Να δούμε τι ιδέες τι πρέπει να αποφύγουμε. Τώρα, μια γενική παρατήρηση για το ότι τελικά δεν πιάνουν τόπο τα, τα μεγάλα πολυφιλόδοξα πρόγραμματα πληροφορικής. Το Eurodac όμω, εγώ ίδιο το δούλεψα, το οποίο παραδόθηκε εγκαίρως και μέσα στον προηγούμενο προπολογισμό, το VIS όχι. Υπήρχε ένα κρατος μέλος που μας καθυστέρησε. Αλλά παρόλα αυτά ήταν στα πλαίσια τα οικονομικά που προβλεπόταν. και το SIS 2 τελικά ε, έφτασε εγκαίρως στα πλαίσια λουπότσων αλλά τελικά δεν ήταν αυτό που περίμενε ο κόσμος. Οπότε ακριβώς και θα πρέπει τα, τα οδυνηρά συμπεράσματα να τα εξαγάγουμε και να φροντίσουμε να πετύχει η πρωτοβουλία αυτή. Να μην κάνουμε λάθη, είπε ο Κιώργο. Μα εντάξει, είναι αναπόφευκτο σε τέτοιε περιπτώσει να υπάρχουν κάποια λάθη αλλά τουλάχιστον να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Κυρία Κέλλερ τώρα. Απαντήσαμε στις επιστολές που μας στείλανε. Έστω και με καθυστέρησε. Μέσα με εβδομάδα άρχισα να ασχολούμαι. Μου είπα να απαντήσω σε όλους τους και οδησυγητές. Οπότε απαντήσεις δόθηκαν και θα δοθούν. Ε, τώρα συμπαθάτε με γι' αυτό το λάθος σχετικά με την 7η Φεβρουαρίου αλλά έχουμε οργανωτικές ε, δυσκολίες, επιμελητίες. Τέλο δεν μπορεί, δεν γινόταν κάτι άλλο. Ε, αυτό είναι το ενακτήριο λάξιμα για τη διαδρομή αυτή. Τεχνικού χαρακτήρα αυτή η συνάντηση τεχνικοί από τα κρατημέλη ε, συζητούν διάφορα τεχνικά στοιχεία. Και αναφέρετε τι έχει κάνει το κάθε κράτος μέλος. Θα η συνάντηση αυτή θα είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει έρχεται. Είστε καλοδεχούμενοι. Ξέρω ότι σας είναι δύσκολο, είστε ίδιοι, αλλά ίσως μπορείτε να στείλετε κάποιο συνεργάτη σας. το μέλλον δεν πρόκειται να οργανώσουμε τέτοιε αντίστοιχε να λάβουμε υπόψη τις υποχρεώσει σα. Για τόσο ο κύριο Κοέλιο ναι ο, το τα του SIS2 αντλήσαμε και από εκεί συμπεράσματα πήραμε μαθήματα είπαμε τώρα, κάνουμε τη μελέτη. Με τη μελέτη θα οριστεί το βεληνικές αυτού του προγράμματος. Δεν μπορώ σήμερα να σας πω ακτιβώς πώς θα είναι το πιλωτικό πρόγραμμα, γιατί τώρα είμαστε στη διαδικασία του να καθορίσουμε το βεληνικές του προγράμματος. Μόλις ε, γίνει η μελέτη, τότε θα ξέρουμε. Πάντως, δεν θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα πρωτότυπο. Θέλουμε να κάνουμε μια δοκιμή τη βάση κάποιων σεναρίων βιομετρικά, χρόνους επεξεργασίας, διάφορα πρακτικά ζητήματα και να δούμε τι είναι εφικτό να γίνει σε ένα πραγματικό ρεαλιστικό περιβάλλον. Άρα πάμε στα κράτη-μέλη, βλέπουμε τι ισχύει και προσπαθούμε στο περιβάλλον αυτό, να συντεριάξουμε αυτό, να προσαρμόσουμε αυτό που θέλουμε να δοκιμαστεί. Οπότε, αυτό μας δίνει ελπίδες ότι αυτό το οποίο θέλουμε να γίνει θα αποδώσει στην πράξη. Μην ξανεχτούμε χωρίς να ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. να ξέρουμε τι θα αποδώσει, τι μπορεί να λειτουργήσει για να μην πρέπει στην διαδρομή κατά την υλοποίηση να αλλάξουμε κάτι. Σας διαβεβαιώ. Δεν έχω συνομιλήσει με καμία απολύτως εταιρεία όσον αφορά αυτό το πακέτο για τα έξυπνα σύνορα. Υπήρχε κάποιος που μας βοηθούσε πριν από χρόνια για τη μελέτη των επιπτώσεων, η Unisys γνωστή εταιρεία. Φυσιολογικό αυτό. Και σε βεβαίω για τις αμερικανικές εταιρείε ότι θα κάνουμε ό,τι προβλέπει ο ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες. Είναι η νομική μας υποχρέωση. Νομίζω ότι σας απάντησα ξεκάθαρα. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα. Όσοι ρωτήσατε. Αν κάτι για την προστασία των δεδομένων και σχετικά δικαιώματα, να πω ότι γνωρίζω, σε μεγάλο βαθμό αυτά έχουν καλυφθεί από τη μελέτη επιπτώσεων. Εάν τώρα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, μεταβολές, γιατί έχει αλλάξει η νομοθεσία, κάτι έχει αλλάξει και ενισχύει τη μελέτη επιπτώσεων, το ξαναδούμε. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι δεν θα συμμορφωθείτε μόνο με τους κανόνες του ΠΟΕ στην εφαρμογή και την κασκαδί του συστήματος, αλλά και με την προστασία δεδομένων που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε λοιπόν στους εισηγητές. Η κυρία Σόμερ, θα αρχίσετε πρώτη. Ή θέλετε να το κάνουμε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την ετοιμότητά της για συνεργασία, ακόμα και αν αυτό δεν μπορεί να συμβεί στις 7 ε, Φεβρουαρίου. Χαίρομαι επίσης ε, ότι αναγνωρίζεται ο ρόλος μας ως ε, συνομοθέτης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο, διότι ξέρω πως δεν είναι για κανέναν, ούτε για το Συμβούλιο, ούτε για το Κοινοβούλιο καλό όταν ε, θεωρούν πως δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ως Τώρα μπορούμε να συμφωνήσουμε για μια εναλλακτική ημερομηνία από τις 7 Φεβρουαρίου για να συζητήσουμε. Θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι η συνεργασία μας με τον ε, κύριο Ένση, τον εισηγητή, ήταν ε, εξαιρετική και είναι εξαιρετική. Όπως επίσης καλή συνεργασία έχουμε και με τους υπόλοιπους κοιόδης εισηγητές. Είναι μια πολύ διάφανη διαδικασία. Και όσον αφορά τα σχόλια του συνάδελφου Κέρκοπ, ότι πρέπει να μην περιοριστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κοιτάξουμε τι γίνεται και πέραν αυτή, για παράδειγμα τα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, πράγματι ε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δίκιο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε 100% την κατάσταση που επικρατεί εκεί με την κατάσταση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως εγώ θα ήμουν πανέτοιμη να ταξιδέψω εκεί στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά. Βέβαια αν, υπάρχει και, ε, αν υπάρχουν και τα κατάλληλα κονδύλια. Και Ίσως μπορέσουμε επίσης πέραν αυτού να δούμε και μία άλλη περίπτωση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ένσιου. Ναι, να σας ενημερώσω ότι ήδη έχω επισκεφθεί τα σύνορα Ενωμένων Πολιτειών Καναδά ως μέλος της ε, αντιπροσωπείας για σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά και χρησιμοποίησα λοιπόν την ευκαιρία αυτή για να επισκεφθώ τα σύνορα αυτά. Να ευχαριστήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πιστεύω ότι τώρα έχουν διευκρινιστεί όλα όσα χρειάζεται να γίνουν και το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεχτεί ότι εμείς θα είμαστε συνομοθέτες και όχι απλοί παρατηρητές είναι ευπρόσδεκτο. Επίσης συμφωνώ με την Πρόεδρο με την ε, απέτησή της από την ε, Επιτροπή να μας δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και την συνεισηγήτρια κυρία Ζόμερ, διότι κατανοεί απόλυτα το στόχο μας, να κάνουμε δηλαδή καλή δουλειά, να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό πακέτο για τα έξυπνα σύνορα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους ε, τους ε, συναδέλφους που συνεργάστηκαν. Είναι ξεκάθαρο ότι το μέλλον των έξυπνων συνόρων είναι αβέβαιο την παρούσα στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, Αβέβαια σύνορα δηλαδή λέει η πρόεδρος. Ωραία συνάδελφοι τότε φτάσαμε στο τέλος αυτής της συνεδρίασης. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την επόμενη 5η 30 Σεπτεμβρίου το πρωί στις 9 και το απόγευμα στις 3. Επόμενη συνεδρίαση 3 Φεβρουαρίου από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στο Στρασβούργο. Κύριε Μπρόνς, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Αν δεν κάνω λάθο και αν κάνω λάθο ε, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, η συνεδρίαση τη 30 ε, Ιανουαρίου δεν προβλεπόταν αρχικά. Εάν όντω ε, ισχύει αυτό, τότε θα ήθελα να πω ότι το να γίνονται συνεδριάσεις που δεν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων είναι μια συνταγή αποτυχίας. Δεν θα έρθει κανείς. η προσέλευση είναι πολύ μικρή και πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να ξοδεύει κανείς 800 λίρες, γιατί τόσο κοστίζει το αεροπορικό εισιτήριο από τον Ηνωμένο Βασίλειο εδώ, για να έρθει και τελικά να μην είναι κανείς. Δυστυχώς ε, θα σας ε, πω και ξέρω ότι θα στεναχωρηθείτε πάρα πολύ, ότι δεν θα είμαι εδώ στις ε, επόμενες ευρώ. δεν θα στεναχωρηθείτε ίσως, το ξέρω. Κυρία Ζόμερ, Μάλιστα να πω λοιπόν και εγώ ότι λυπάμαι πάρα πολύ για το ότι αυξάνεται η συχνότητα συνεδριάσεων στο Στραμβούργο Και να τονίσω ότι δεν πρέπει αυτό να γίνει συνήθεια. Κανονικά δεν πρέπει να γίνονται συνεδριάσεις επιτροπών στο Στρασβούργο εκτός από έκτακτες περιπτώσεις. Και πραγματικά θα ήθελα να δηλώσω την ε, απογοήτευσή μου για αυτό το φαινόμενο που ολοένα και εντείνεται. Συμφωνώ και με τους δύο. Νομίζω πως έχουμε περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων της Επιτροπής αυτής, διότι ολόνα και προστίθενται συνεδριάσεις σε ένα ήδη φορτωμένο πρόγραμμα και πραγματικά θα αποτρελαθούμε από το φόρτο εργασίας και τη συχνότητα των συνεδριάσεων. Και η αλήθεια είναι ότι τις συνεδριάσεις που ήδη έχουμε δεν τις χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν τις αξιοποιούμε. Και προσωπικά με κατακλείζουν email για αλλαγή στο πρόγραμμα, για συνεδριάσεις που, ακυριάσεις που αναβάλλονται, που ε, παρατείνονται, συντομεύουν και τα χάνω. Σήμερα είχα την εντύπωση, για παράδειγμα, ότι η συνεδρίαση θα άρχισε στις 9 και άρχισε 10 παρατέταρτο και ήταν σίγουρα σε ένα από τα 35 email που πήρα σήμερα το πρωί σχετικά, αλλά αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να ε, μεταφέρουμε στην Γραμματεία και στον Πρόεδρο να μας ε, επιτρέψει να προγραμματίσουμε καλύτερα τον κύκλο εργασιών μας. Σας ευχαριστώ όπως και να έχει. Ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε πολύ τους διερμηνείς. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.